Καλησπέρα σας. Μπορούμε να ε, σας πω ότι υπάρχουν τα κείμενα που υιοθετήθηκαν χθες, τα πρακτικά είναι στη διάθεσή σας, υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν βλέπω να έχει κανένας καμία παρατηρήση. Εγκρίνω λοιπόν τα πρακτικά αυτά. Προτού τώρα